Welcome Καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μανουέλ Μπαρόσο. Θα ήθελα να σας πω ότι ακολουθεί σύμφωνα με τη Μέση Διάταξη δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 7 Μαΐου. Θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στον Υπουργό κύριο Λόπε Καρίδα, εξ του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, στις 7 του μηνός, αυτή τη βδομάδα δηλαδή ακόμα, υπάρχει συνεδρίαση των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. και γι' αυτό συζητάμε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη τόσο σημαντική συνάντηση που έχει ως αντικείμενο να επισημοποιήσει την ε, συμφωνία η οποία επιτεύχθη για δανειοδότηση προς την Ελλάδα, το πακέτο δηλαδή οικονομικής στήριξης στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί η σοβαρή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αυτής της Ευρωζώνης. Επίσης, η συνάντηση αυτή θα εξετάσει και θα προβληματιστεί σε σχέση με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε από αυτήν την κατάσταση, από τη συμφωνία για το μέλλον της Ευρωζώνης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων αυτό που θα κάνουν την Παρασκευή είναι ότι θα επιβεβαιώσουν την οικονομική λύση που βρέθηκε για την Ελλάδα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα επισημοποιήσουν την δέσμευση, πολιτική δέσμευση καταρχήν, που ανελήφθη ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου από τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, δέσμευση προς την Ελλάδα, αλληλεγγύης, προκειμένου να μπορέσει να λύσει την τόσο δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει. Οπότε, την Παρασκευή, οι ηγέτες κατόκια κυβερνήσεων θα υποβάλουν, θα παρουσιάσουν, θα συμφωνήσουν για την διαθεσιμότητα των 15 υπολείπων μελών της Ευρωζώνης, ώστε άπαξ και η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, οικονομικών προσαρμογών, η χώρα αυτή θα μπορέσει να πάρει τα χρήματα που αποφασίστηκαν με στόχο την σταθερότητα και ολόκληρης της Ευρωζώνης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, αποφασίστηκε ως πολιτική δέσμευση ήδη στις 11 Φεβρουαρίου από τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Αυτή η απόφαση είναι σημαντική και είναι και πολιτικά πολύ σημαντική και ιστορικά πολύ σημαντική, διότι πρόκειται για μια αναγκαία απόφαση για την αξιοπιστία της Ευρωζώνης. Για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, προς τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σημαντική επίσης για την ε, καλή κατάσταση των δημοσιονομικών, κάτι το οποίο απαιτεί η ίδια η δημιουργία της Ευρωζώνης. Και είναι επίσης μια πολύ σημαντική απόφαση προκειμένου να έχουμε μια πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο Επίτροπος Όλη Ρεν, παρόν εδώ, έκανε γνωστές τις αποφάσεις για την περίοδο μέχρι το 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως μήνυμα έχει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μετά από την χειρότερη ύφεση της ιστορίας της προβλέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να αναπτυχθεί με 1% το 2010 και 1,75% το 2011. Συνεπώς, η οικονομική ύφεση έληξε και ξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη στην οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολύ το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης και αποφάσεις των κρατών μελών να δώσουν πολύ σημαντικά ποσά στην οικονομία προερχόμενα από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών αλλά και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχοντας περάσει από τη χειρότερη, επαναλαμβάνω, χειρότερη περίοδο ύφεση στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη σε ανάκαμψη. Αυτές είναι οι προβλέψεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίχως άλλο, η απόφαση για την Ελλάδα η απόφαση των δανείων προς την Ελλάδα συνεισφέρει αποφασιστικά για την πραγματοποίηση της ανάκαμψης, της βιώσιμης ανάκαμψης στην Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε σωστά στη σημερινή κατάσταση έκανε ό,τι μπορούσε για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την πάρα πολύ σοβαρή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί τελικά αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς τους τελευταίους μήνες είναι ότι έκανε ξεκάθαρα βήματα προς την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε ξεκάθαρα βήματα τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να φάνηκαν ότι πάνε πάρα πολύ αργά. Όμως γίνανε βήματα με ασφάλεια και αποφασιστικότητα. Και θα καταλήξουν την Παρασκευή που μας έρχεται στην επιβεβαίωση αυτή από πλευρά των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων. Εμείς θέλουμε η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στέρες βάσεις. Πρώτον, υπευθυνότητα υπευθυνότητα σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Όταν υπογράφεται μια συνθήκη, να προχωράει. Δεύτερον, επίδειξη αλληλεγγύης. Αυτή είναι μια αρχή που βρίσκεται στην ίδια την ψυχή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, συντονισμός. Συντονισμός για τα δημοσιονομικά και για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, στους 20 για παράδειγμα, και επίσης για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι το έγγραφο που ετοιμάζει ο Επίτροπος Όλη Ρεν και που θα υποβληθεί στις 12 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θέλω να πω ότι μια οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν αυτή που ετοιμάζεται τώρα βάζει βάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αποτελεσματικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εποπτεία και είμαι πεπισμένος ότι θα αναφέρεται σε αυτό το άγγραφο που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έλεγχος λοιπόν των δημοσιονομικών και εποπτεία των οικονομικών συστημάτων στην Ευρώπη. Θα έκανε έκκληση λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα το πακέτο δημοσιονομικής εποπτείας που συζητιέται αυτή την εποχή εδώ σε εσά τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Χρειάζονται επίσης μηχανισμοί πρόληψης για να προλάβουμε νέες κρίσεις. Και τέλος, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή όταν εκπροσωπείται προς τα έξω. Στους 20, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι βήματα προς μια καλή οικονομική διακυβέρνηση. Ο δανεισμός προς την Ελλάδα είναι ένα κομμάτι όλου αυτού του συνόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σίγουρος, πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτήν επέλεξε και είμαι πεπισμένος ότι οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων θα εγκρίνουν αυτό το πακέτο δημοσιονομικής στήριξης προς την Ελλάδα που αποτελεί, όπως είπανε και στις 11 Φεβρουαρίου οι ίδιοι οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων που θα βοηθήσει γενικότερα τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Μου ζητήθηκε να κάνω μια δήλωση προς το σώμα πριν από την διάσκεψη της Ευρωζώνης. Καταρχήν να εκφράσω τη συλληπιτήριά μου για τις οικογένειες των θυμάτων στην Αθήνα σήμερα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βία. Να σας ανακοινώσω το πακέτο για την Ελλάδα που εγκρίθηκε την περασμένη Κυριακή και θα σας δώσω κάποιες από τις απόψεις μου όσον αφορά την αποφυγή νέων κρίσεων τέτοιου τύπου. Όσον αφορά την Ελλάδα, ένα πολυετές πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης συμφωνήθηκε με τις ελληνικές αρχές. Αυτό από κοινού προετοιμάστηκε με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε ένα σταθερό και συμπαγές και αποξιόπιστο πακέτο που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα οδηγήσει στην ανάκαμψη. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ε, το θάρρος που έδειξε ο, Πρωθυπουργό ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Σε αντάλλαγμα, σύσταση της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο συντονισμένος ευρωπαϊκός μηχανισμός για την βοήθεια στην Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί και είναι μια ανευπρεγουμένου ενέργεια αλληλεγγύης που δεν έχει το αντίστοιχό της σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποφασίστηκε λοιπόν να βοηθηθεί η Ελλάδα για να επανέλθει στην σωστή πορεία η Ελλάδα και να προστατευτεί και ολόκληρη η Ευρωζώνη. Ε, η Κομισιόν θέλει να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενώ βασίζεται σε διμερείς, ε, διμερή δάνεια είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Η Κομισιόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του και στη, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και την εφαρμογή του. Η Κομισιόν θα παραμείνει κεντρικός άξονας αξιολόγησης του, της απόδοσης της Ελλάδας ε, γιατί θα ελέγχει και θα υποπτεύει την τήρηση των όρων. Μέχρι το τέλο τη εβδομάδα θα έχουμε μια κρίσιμη μάζα 100 μελών που ήδη θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε να παρέχουν αυτά τα διμερή δάνεια στην Ελλάδα. Είναι δική μου πεποίθηση ότι η άνευ οικονομική στήριξη προς την Ελλάδα, 110 δις ευρώ, και το πρόγραμμα προσαρμογής είναι η κατάλληλη απάντηση για την ελληνική κρίση. Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε πως σταθερά θα εφαρμοστεί και από την Ελλάδα και από τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης. Αυτή την άποψη έχουν και άλλοι. Όπως για παράδειγμα διαπίστωσα υποστηρικτικές δηλώσεις για τις τις ε, του πρώην ε, τρέχοντος και μελλοντικού προέδρου της, του G20. Για όσους δεν είναι απόλυτα πεπισμένοι θα πρέπει να τους πούμε πως κάνουν λάθος και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Στην διάσκεψη τώρα των ε, μελών της Ευρωζώνης την Παρασκευή θα εξετάσουμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αποκομίσουμε τα σωστά διδάγματα από αυτή την κατάσταση. Η συζήτηση φυσικά θα αποτελέσει ένα σημείο κίνησης, διότι οι αποφάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται και θα αναλαμβληθούν με όλα τα 27 κράτη-μέλη, όσους είναι δηλαδή μέλη της Ευρωζώνης και όσους όχι. Και θα πρέπει σαφώς να δηλώσω πως η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο των 27 είναι μια πηγή δύναμης. Ενώ πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας, ε, το γεγονός είναι ότι η κοινή δράση των 27 που δεν έχει το, το αντίστοιχο της ολόκληρο τον κόσμο δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να προβληματιστούμε και να ενεργήσουμε για τα εξή. Καταρχήν, κανόνα οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερον, μεταρρύθμιση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Η Κομισιόν εργάζεται εντατικά για την οικονομική διακυβέρνηση και είναι έτοιμη να παρουσιάσει τι προτάσει τη για το πώ θα βελτιωθεί αυτή την επόμενη Τετάρτη. Υπάρχουν τρία, βασικά, βασικοί άξονε που πρέπει να εξεταστούν. Καταρχήν, ευθύνη. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή και τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Δεύτερον, ε, η επιβολή της πρόληψης αλλά και ε, της πρόληψης στο πακέτο αυτό είναι πολύ σημαντική. Τώρα, ακόμη και όσοι αμφισβητούσαν την ύπαρξη ενό συμφώνου τέτοιου, τώρα είναι υπέρ αυστηρότερων κανόνων και αυστηρή εφαρμογή του. Δεύτερον, αλληλεξάρτηση. Όλοι μαζί είμαστε στο ίδιο καράβι. Νομίζω πως η κρίση αυτή έχει δείξει σαφώ πως η έλλειψη ισορροπίας, οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωζώνη ιδιαίτερα, ε, δείχνει αποκλήσεις και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που οδηγεί σε άλλου είδους ε, ανισορροπίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένοι θα πρέπει να είναι μία ανταγωνιστική ώστε οι άλλοι φαίνονται σχετικά πιο ανταγωνιστικοί. Όλοι μας ανταγωνιζόμαστε στην ίδια παγκόσμια αγορά. Αυτό που χρειάζεται είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με έναν ισόρροπο και αμοιβαία ενισχυτικό τρόπο. Πιστεύω πως ε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για ανισορροπία. Γι' αυτό θα προτείνουμε αυξημένη εποπτεία και αυξημένο συντονισμό οικονομικής, οικονομικών πολιτικών. Είμαι ευτυχής που τώρα βλέπω μεγαλύτερο άνοιγμα όσον αφορά τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. We Να... Επίσης να ολοκληρώσουμε ένα σύστημα οικονομικών κανόνων, έναν μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, δύσκολες καταστάσεις. Καλύτερα είναι να είμαστε ασφαλείς παρά μετά να πληρώνουμε τα σπασμένα. Πιστεύω ότι από πολιτικής άποψης και όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, βρισκόμαστε, διανύουμε μια περίοδο όπου αν δεν κάνουμε ένα σημαντικό άλμο θα μείνουμε πίσω. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, η στιγμή που ζούμε αυτή τη ε, σήμερα στην Ευρώπη, όπου η αλληλεγγύη μας, η ευθύνη μας δοκιμάζονται καθημερινά. Ελπίζω πως οι ηγέτες των κρατών μελών μας θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όχι μόνο για να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά για να δείξουν την ευθύνη τους, την υπευθυνότητά τους και την αφοσίωσή τους στο κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, θα πρέπει να γίνουν στη βάση ε, αδιαμφισβήτητων αλλαγών που ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα πρέπει να γίνουν πιο αποφασιστικά και γρηγορότερα από ό,τι αρχικά είχαμε υπολογίσει πριν την κρίση. Θα πρέπει ωστόσο επίση να πούμε πω δεν μπορούμε να γνωρούμε το γεγονό ότι η δημοσιονομική επιδείνωση του 2009 βασικά οφείλεται στην λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών εν ώψη άνευ πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας που οφειλόταν σε παράγοντες εκτός Ευρώπης. Τα προβλήματα στην Ευρωζώνη ήταν βασικά αποτελέσματα πολιτικών κατά της ύφεσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, έπρεπε η δική μα πολιτική να διορθώνεται κάθε φορά και τα κράτη-μέλη έπρεπε να προβούν σε μεταρρυθμίσει, Για παράδειγμα, του συνταξιδοτικού του συστήματο, Η ευθύνη των κυβερνήσεων θα πρέπει να συμβαδίζει με την πορεία τη δημοσιο... της χρηματοπιστωτικής και γι' αυτό και θα πρέπει να υποστηρίξουμε έναν χρηματοπιστωτικό τομέα υπεύθυνο και αποτελεσματικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πω οι χρηματοπιστωτικές αγορέ είναι, μάλλον οι τη χρηματοπιστωτική είναι πολύ σημαντικοί για να καθοδηγήσουμε οδηγήσουν την αίσθηση των αγορών, των χρηματαγορών. Η έλλειψη ευθύνη είναι που οδήγησε στην κρίση και ε, γι' αυτό και χρειαζόμαστε πολύ ισχυρότερε ε, χρηματαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουμε τι επενδύσει για τη μελλοντική ανάπτυξη σύμφωνα με το όραμα για το 2020. Θα πρέπει να έχουμε υπεύθυνη ανταπόκριση από όλου του φορεί τη αγορά. Ήδη έχουμε κάνει πολλά όσον αφορά την μεταρρύθμιση των ε, χρηματαγορών και βασίζομαι σε εσά ώστε αυτό να καταστεί σαφέ σε όλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει και θα πρέπει να, θεωρηθεί, να, να φαίνεται πω ενεργεί από κοινού Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Κομισιόν. Πιο ασφαλείς αγορές παραγόγων, καλύτερη εποπτεία των χρηματαγορών, διασφάλιση πως οι, οι, οι τράπεζες έχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να καλύπτουν τους, ίδιου τους ίδιους κινδύνους τους ε, δεν έχουν ήδη ξεκινήσει οι μεταρρυθμίσει. Όπω είπα πριν από δύο εβδομάδε στο Σώμα, ελπίζω πω γρήγορα θα υπάρξει πρόοδο στην πρότασή μα για τα ε, hedge funds και τα private equity. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Συστημικό Κίνδυνο που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2011. Αλλά δεν μείνουν όλα αυτά στα χαρτιά μόνο. Ε, ε, θα πρέπει να έχουν και τα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Δηλαδή, τέτοιες εξουσίες που θα μπορούν να επιβάλλουν ευρωπαϊκούς κανόνες και επιμένω σε αυτό, ευρωπαϊκούς κανόνες, όχι μόνο εθνικούς κανόνες, και να ρυθμίζουν οποιαδήποτε διαφορά μέσα στο πλαίσιο του συνόλου των διεθνών εποπτών. Ε, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να ληφθούν και να είναι και φιλόδοξες. Και άλλες προτάσεις θα γίνουν φέτος για να βελτιωθούν η βελτιωθεί η προστασία του καταθέτη και του επενδυτή, να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα του τραπεζικού κεφαλαίου και να αποκλειστεί η υπερβολική μόχλευση. Τους τελευταίους μήνες και ακόμα και αυτό το μήνα η κατάσταση στις αγορές ε, κρατικού χρέους έχει ε, ξεφύγει. Σε κάποιες χώρες ε, υπήρξε πρόταση ε, για νομοθεσία για να, να τυποποιηθούν τα παράγωγα, να υπάρξει σωστή εποπτεία και ρύθμιση. Και τώρα εξετάζουμε αν χρειάζονται περαιτέρω ειδικά μέτρα όσον αφορά τα παράγωγα που αφορούν το κρατικό χρέος. Αυτοί οι φορεί τώρα αξιολόγησης, επιστοληπτικής ικανότητα είναι επίση πολύ σημαντική για την αγορά, αλλά θα πρέπει να βασίζονται σε γενικές κινήσεις αγοράς και όχι, και όχι, τη, και όχι στις βασικές, στα βασικά στοιχεία. Γιατί αυτέ οι, οι οργανισμοί έχουν τόσο μεγάλο ρόλο και επιρροή στην αγορά, έχουν ωστόσο ταυτόχρονα την ευθύνη να διασφαλίζουν πω οι αξιολογήσεις του είναι... Ε, βάσιμες ε, και κατανοητές και γι' αυτό και προτείναμε νέα νομοθεσία για αυτές τις, ε, αυτούς τους οργανισμούς που θα αρχίσει να ισχύει στους επόμενους μήνες ώστε να διασφαλίσουμε πως οι οργανισμοί αξιο ε, αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα λειτουργούν υπεύθυνα πιστεύουμε πως θα πρέπει να τεθούν υπό την άμεση υποπτία της ε, μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Χρεογράφων. Σκεφτόμαστε επίσης μήπως χρειάζονται μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή αξιολόγηση του κρατικού χρέου πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει να βάλουμε τάξη στα του οίκου μα, ενώ θα, θα, θα παροτρύνουμε και τους υπολείπους να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή οι χρηματαγορές, οι ασφαλιστικέ αγορές δεν είναι παιδική χαρά για τους ε, κερδοσκόπου. Η ελεύθερη αγορά σημαίνει κανόνες και συμμόρφωση προς αυτούς ώστε να ξέρει ο καθένας τι δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και τι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πρέπει να, υπηρεσίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ακριβώς αυτό, μια υπηρεσία και όχι αυτός σκοπός, θα πρέπει να είναι αποσπασμένες από την λειτουργία τους. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί τελικά οι φορολογούμενοι σταθεροποιούν τις αγορές σε περιπτώσεις χρηματοπιστωτικής κρίση και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα για το μέλλον και το μήνυμα για αυτή την Παρασκευή στην Ευρωζώνη θα είναι σαφές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε όλα τα μέτωπα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα ε, θα θέλαμε και εμείς να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας ε, προς τις οικογένειες των θυμάτων στην Αθήνα που μας αναφέρατε ότι έγιναν επεισόδια. Ελπίζουμε το αδιέξοδο αυτό στην Ελλάδα να τερματιστεί προς όφελος όλων μας. Και τώρα ακολουθούν οι αγορητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο έχει ο Ζωζεφ Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη ζούμε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Με τη σοβαρή κρίση στην Ελλάδα, τις συνέπειές της στους πολίτες και μόλις το θυμήσατε κι εσείς, τραγικές συνέπειες, δραματικές συνέπειες αυξάνονται τα ελλείμματα στα περισσότερα κράτη-μέλη μας. Ευρωπαϊκή ανταπόκριση που δεν είναι πάντα στο ύψος των προσδοκιών μας. Αλλά με ευρωπαϊκή ε, απάντηση που ε, αν μη τι άλλο υπάρχει. Σήμερα έχει έρθει η ώρα οι Ευρωπαίοι να βγάλουν τα διδάγματα από ε, τα γεγονότα αυτά και να κάνουν σημαντική και βαθιά μεταρρύθμιση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Για να σταματήσουν να αποφασίζουν μόνα τους τα κράτη-μέλη χωρίς συνεννόηση με τους εταίρους τους που κατά τα άλλα έχουν κοινό νόμισμα και κοινέ αξίες. Ε, ε, μια κοινή μοίρα. Δεν μπορούν λοιπόν να αποφασίζουν μόνοι τους για τις προτεραιότητες δημοσιονομικές, κοινωνικές και φορολογικέ. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και στι νοοτροπίες, έτσι ώστε τα κόμματά μας, οι υπουργοί μας, τα εθνικά σώματα να σταματήσουν συστηματικά να μειώνουν, να υπονομεύουν ό,τι αποφασίζεται στην Ευρώπη. Ενώ οι ίδιοι συμμετέχουν στις αποφάσεις αυτές. Μα πώς είναι δυνατόν ακόμα για μεγάλο χρονικό διάστημα να επικαλούμαστε την αλληλεγγύη των εταίρων μας όταν είμαστε σε δύσκολη θέση και να τους αγνοούμε πανηγυρικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όταν επανέρχεται η τάξη. Επιτρέπεται ακόμα να ζητούμε σημαντική βοήθεια από τους εταίρους μας χωρίς να μπορούμε να εγγυούμεθα τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στους ε, ε, δημοσίου λογαριασμούς. Είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να εκπλησόμαστε που αυτά τα θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια όταν επικαλούμαστε στην αλληλεγγύη των λαών, αλλά υπάρχουν κάποιοι λαοί που δουλεύουν 35 ώρες την εβδομάδα και βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 60, ενώ άλλοι 48 και άνω και βγαίνουν στη σύνταξη στα 67 έτη. Ε, δεν γίνεται αυτό. Ε, το αντίθετο ε, πιστεύω, ότι έχει έρθει η ώρα να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα και να δώσουμε σωστές απαντήσεις ε, και τις αληθινές που δεν είναι εθνικές αλλά ευρωπαϊκές στο σημερινό κόσμο. Οι απαντήσεις αυτές δεν είναι της τάξης της δημαγωγίας αλλά της ευθύνης και ε, του κοινού νου. Τις απαντήσεις αυτές θα πρέπει εμείς να τις δώσουμε χωρίς ολιγορία. Γιατί αν δεν το πράξουμε θα επιβληθούν σε μας πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Και δεν θα μας κατηγορήσουν και εύγολα, εύλογα οι λαοί μας ότι δεν κάναμε το καθήκον μας, ότι τους είπαμε ψέματα, αλλά επιπλέον θα αναγκαστούν να δεχθούν πολύ πιο σημαντικές ε, αποφάσεις από αυτές που καλούμαστε σήμερα να πάρουμε. Θα πρέπει με τρόπο ξεκάθαρο να ζητήσουμε μια Ευρώπη οικονομική, κοινωνική και φορολογική. Γι' αυτό χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα από πλευράς των κυβερνησεών μας, δεξιών και αριστερών θα τα ακούσει αυτά το Συμβούλιο που λέμε. Θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε να ακούσει. Με, το ρωτάω τον Κίφερ Χόφστατ εδώ που ε, έχει ζήσει το Συμβούλιο. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει, να συζητήσει στο Συμβούλιο. Αυτό το λόγο μας τον ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελπίζω. Και αγαπητέ Ζωζέ Μανουέλ, σας ε, καλώ ε, να το πράξετε και ως θεματοφύλακα της συνθήκη, να επαγρυπνείτε ώστε οι αποφάσεις που παίρνουμε να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, διαπιστώνω ότι για την ε, ε, οδηγία για τις υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται και χάνουμε χρήματα και χάνουμε και ανάπτυξη. Δεν επιτρέπεται πια αυτό. Δεν είμαι ουτοπικός, ούτε και αφελής πιστεύω κυρίες και κύριοι, αλλά έχει έρθει η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Και σας προτείνω αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουμε με θάρρος, σθένο με αίσθημα ευθύνη όπω έκαναν πριν από 60 χρόνια οι πατέρε τη Ευρώπη, Σούμαν, Ντεγκάσπαρη, Αντενάουερ κλπ. Οι πατέρες τη Ευρώπη που δεν δίστασαν να πάρουν θαραλέες αποφάσει, εμπνευσμένε, με όραμα. Θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Δεν κάνανε δημοψηφίσματα με ολιγορίε και καθυστερήσει. Ε, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους με πολιτικό σθένος και απάντησαν στις επιταγές των καιρών. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί η κρίση που ζούμε να αποδειχτεί σωτήρια. Αν έχουμε το θάρρος να λάβουμε τα, καλά, τα σωστά μέτρα, αλλά μπορεί να είναι και ολέθρια εάν ε, χάσουμε την ευκαιρία αυτή για τις μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται επιγόντως οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση στην Ευρώπη, προσαρμογή των φορολογικών κανόνων. Και τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε τεχνητό χάσμα ανάμεσα στις χώρες μέλη του ευρώ και στις άλλες. Η αλληλεγγύη ισχύει και για τα 27 μέλη. Και σας το ζητώ, κύριοι υπεύθυνοι του Συμβουλίου. Κοιτάξτε την Ευρώπη κατάματα. Σας ζητώ, κάντε τις μελέτες υπολογίστε τι θα συμβεί αν αύριο η Γαλλία και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με την Ελλάδα. Πού θα πάει το ευρώ μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όλοι μαζί έχουμε αυτή την κοινή ευθύνη αυτή τη στιγμή και ο χρόνος δεν περιμένει. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, ένας από τους συναδέλφους Μαρή Ματλέν έχει ζητήσει το λόγο με την μπλε κάρτα. Εγώ δεν σας έχω στον κατάλογο μιλητών όμως. Μπαρή Ματλέν, σε μερικά λεπτά θα σας δώσω το λόγο. Θα πάρετε το λόγο, ναι, τώρα σας βλέπω εδώ. Τώρα, εκ, μέλους, μέρους των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μπάντια Κουτζέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μα προ τον ελληνικό λαό για του θανάτου που έλαβαν χώρα σήμερα. Και θέλω επίση να κάνω μια έκκληση για να επιστρέψει η ηρεμία. Εμεί στηρίζουμε του Έλληνε, έχουν την αλληλεγγύη μα στην προσπάθεια που κάνουν μέσα σε μια μακρά διαδικασία. Θέλω επίσης να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και να τον ενθαρρύνω στο πολιτικό του θάρρος προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα και να έχει ένα καλό μέλλον η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουμε ότι θα συνοδεύσει τις διαδικασίες μεταρρύθμισης που είναι αναγκαίες. Δεν είναι δυνατόν να αρκεστούμε σε έναν απλό έλεγχο από πλευρά μα πρέπει να αποτελέσουμε μέρο τη μεταρρύθμιση, να τη συνοδεύσουμε. Η επιτυχία τροποποίηση θα πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια και μια κοινή επιτυχία μια ενωμένη Ευρώπη που έχει κοινό μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα πολιτικά μέσα από την Ευρώπη και τα φορολογικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Να δώσουμε ό,τι βοήθεια αρρωγή χρειάζεται σε αυτό το δύσκολο στάδιο. Πέρα από την ελληνική κρίση όμως πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ε, ιδιαίτερα ταραγμένες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα που έχουμε πάρει από το παρελθόν για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και να φτιάξουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην είναι μόνο νομισματική αλλά και πραγματικά οικονομική. Η εποχή του Ζακ ε, Ντελόρ πέρασε, τώρα πρέπει να περάσουμε σε άλλα πράγματα, αυτά που απαιτούν οι εποχέ. Για να πετύχουμε αυτού του στόχου, του τόσο φιλόδοξου, πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μα. Το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη είναι μία από, ένα από τα πράγματα τα οποία έδειξαν ότι είναι αναγκαίο ο συντονισμό των οικονομικών μα πολιτικών. Ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών πρέπει να προχωρήσει και να μας πάει σε μία αηφόρο ισχυρή ανάπτυξη που, από την οποία να χαίρουν όλοι και θέσει εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα κάνει τολμηρέ προτάσει από αυτού που θα ξεπερνάν την απλή λογική της καταστολής. Πρέπει να μάθουμε να χτίζουμε και μαζί να ενισχυθούμε περισσότερο. Ελπίζω, Πρόεδρε Μπαρόσο, να αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσετε τον ρόλο σας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έπακρο. Επίσης, χρειαζόμαστε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Οικονομική Σταθερότητα. Είναι μια πρόταση που ήδη από τον Μάρτιο ενέκριναν οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων. Δεν πρέπει να έχουμε και να επιτρέπουμε την κερδοσκοπική συμπεριφορά. Πρέπει να έχουμε σχεδιασμό για έναν μηχανισμό που θα μας βγάζει από κρίσεις. Πρέπει επίσης να αναπτύξουμε και μια νέα έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Έχουμε κοινό προορισμό ή αλλιώς καταδικαζόμαστε σε μια αρνητική δυναμική από τους εθνικούς εγωισμούς και από την καταστροφική διάθεση μεταξύ μας. Πρέπει να μάθουμε ότι θα μείνουμε και θα ζήσουμε μαζί. Η σημερινή κρίση αποτελεί μια δοκιμή για μας. Έπειτα, ο οικονομικό χώρο πρέπει να πάρει τι διαστάσει που του πρέπει. Του επόμενου μήνε και εβδομάδε έχουμε την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει θέση για διάφορε νομοθετικέ προτάσει πάρα πολύ σημαντικέ, όπως είναι τα Ταμεία οικονομική κάλυψη, η Οικονομική Εποπτεία. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τα θεσμικά όργανα να μα στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή, ώστε να διασφαλίσουμε η Ευρώπη πολύ γρήγορα να έχει ένα σύστημα ρύθμισης και εποπτείας. Ελπίζουμε οι κοινέ αυτές προσπάθειες θα οδηγήσουν και στη δημιουργία ενός φόρου για τις οικονομικές συναλλαγές με στόχο να συμμετάσχουν όλοι αναλογικά στην οικονομική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι. Το μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη και από την ε, ενίσχυση τη δικιά μας που είμαστε κύριε εταίροι της. Αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά με τη στρατηγική 2020, αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε περιεχόμενο σε μια κοινή πολιτική ατζέντα και αν καταδικάσουμε τις οικονομίες μας σε μια χαμηλή ανάπτυξη με ελάχιστε ευκαιρίε απασχόλησης, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να αποφύγουμε νέες επιθέσεις οι οποίες θα είναι πιο σοβαρές και που πιο δύσκολα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Το μέλλον τη Υπήρου μα διακυδεύεται εδώ. Από τη δικιά μα ευφυα και τη δικιά μα ελληνική, από τη δικιά μα αποφασιστικότητα εξαρτάται το μέλλον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Γκίφερ Χόφστατ, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, πρόεδρος. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή ότι και εκφράζω εδώ όλου του συναδέλφου και τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ο μηχανισμό αυτό που δημιουργήσαμε θα λειτουργήσει. Από την αρχή είχα τις επιφυλάξεις μου και τις επικρίσεις μου για το μηχανισμό αυτό των διμερών δανείων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ελπίζω ότι θα λειτουργήσει το σύστημα, επειδή είχα επιφυλάξεις για να τερματίσει τη ε, κερδοσκοπία εις βάρος του ευρώ. Γιατί σιγά σιγά αγαπητοί συνάδελφοι περί αυτού πρόκειται. Κερδοσκοπία και απειλή κατά του ευρώ. Δεν επιτίθενται ε, στην Ελλάδα απλώς ή όπου ε, αφορά τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Είναι πολύ ευρύτερο και πολύ σοβαρότερο αυτό που συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή τώρα επισημοποιηθεί στις 7 του μηνός ο μηχανισμός αυτός, ελπίζω να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως. Για το μοναδικό λόγο ότι δεν έχουμε άλλο μέσο στη διάθεσή μας. Δεν θέτουμε άλλο εργαλείο. Θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό και να υποστηρίξουμε το μηχανισμό αυτό. Αλλά, και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο μου, θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης πολύ καλά ότι στο προσεχές μέλλον δεν θα μπορούμε κάθε φορά να χρησιμοποιούμε αυτό το μηχανισμό. Έτσι, θα πρέπει να βρούμε ένα διαρθρωτικό μηχανισμό μηχανισμό το συντομότερο. Όχι του επόμενου μήνε, σας ελπίσουμε να χρειαστεί, αλλά για τα επόμενα έτη αν μη τι άλλο, γιατί θα ξαναζήσουμε τέτοιε καταστάσει. Και αν θέλουμε να έχουμε διαρθρωτικό μηχανισμό για το μέλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το εξή. Θα πρέπει να βγάλουμε τα ε, διδάγματα από τις εξελίξεις των τελευταίων πέντε μηνών. Πέντε μήνες χρειαστήκαμε για να βάλουμε ένα μηχανισμό σε θέση. Τρεις μήνες για να αποφασίσουμε επί της αρχής και δύο μήνες για τις λεπτομέρειες και τους όρους. Γιατί, Γιατί το σύστημα είναι διακυβερνητικό. Ε, ε, για άλλη μια φορά λέγω και πιστεύω ότι το πρώτο δίδαγμα που πρέπει να εξάγουμε για το μέλλον είναι ότι ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κοινοτική της προσέγγιση γιατί είχε προτείνει από την αρχή ε, Ευρωπαϊκό Δάνειο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε αποφασίσει αμέσως το Δεκέμβριο είναι το Γενάρη και ήδη να αποδίδει οπότε ε, θα σταματούσαν αυτές οι κερδοσκοπικές κινήσεις κατά του ευρώ. Ελπίζω στις 7 του μηνός η πρώτη απόφαση που θα ληφθεί και το πρώτο μάθημα που θα βγάλουν από τους 5 είναι να πούνε ότι εντάξει α ελπίσουμε τώρα αυτό να λειτουργήσει αλλά ει το εξή θα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει πρόταση ε, για ένα κοινοτικό δάνειο που να μπορεί να αποφασίζεται αμέσω για να σταματάει μαχαίρι η κερδοσκοπία ε, απέναντι στο ευρώ. Γιατί όλη η ρευστότητα και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται και, βρίσκεται πίσω από ένα τέτοιο δάνειο. Ενώ στο διακυβερνητικό χρειάζονται 16 χώρε να δώσουν το OK, ίσως και 16 κοινοβούλια μετά. Εντάξει, ξέρω ότι ο κύριο Όλη Ρεν έχει αρχίσει να κάνει ήδη προτάσει και το δεύτερο λοιπόν δίδαγμα είναι ότι χρειάζονται διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο πρόληψης στο σχέδιο σταθερότητας, στο σύμφωνο σταθερότητας, ένα ευρωπαϊκό ας πούμε, νομισματικό ταμείο, ένα διαρθρωτικό μηχανισμό, στον οποίο να ανατρέχουμε αμέσως και ένα τρίτο μια στρατηγική για το 2020 που είναι πολύ πιο στιβαρή από αυτή που έχουμε σήμερα επιτάπητος και συζητούμε. Και κάτι άλλο επίσης για τους οίκους αυτούς αξιολόγησης ή βαθμονόμησης. Ε, ξέρουμε ότι είναι σαν τον καιρό της προγνώσης. Όταν ε, είναι πολύ σκληρές, πολύ αυστηρές, τις θέλουμε πιο χαλαρές. Όταν είναι χαλαρές, θέλουμε πιο αυστηρές. Εν περιπτώσει. Πάντως, αυτή η κοινοτική μέθοδος είναι μια καλή ε, λύση και θα πρέπει να την εξετάσουμε. Και τέλος, Πρόεδρε, έκκληση στην Ισπανική Προεδρία να εγκρίνει την ε, εποπτεία των χρηματοοικονομικών. Ζητώ συγγνώμη κύριε Υπουργέ, δεν φταίμε εμεί. φταίει το Συμβούλιο που άλλαξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι δεν είναι. Είχε κάνει πρόταση η Επιτροπή, της οποίας είχα επικρίνει, αλλά ήταν πολύ πιο πέρα από αυτό που έκανε το Συμβούλιο. Και τώρα εμείς ξανακάνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω να σας κάνω μια καλή πρόταση. Εάν θέλετε η ε, χρηματοοικονομική εποπτεία και οι ρυθμίσεις να εφαρμοστούν σε ένα μήνα, δεχτείτε αμέσως στο Συμβούλιο και στο ΕΚΟΦΗΝ τις τροπολογίες που θα σας κάνει το Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Πολύ εύκολο και γρήγορο αυτό να γίνει για τη χρηματοοικονομική εποπτεία να αρχίσει να ισχύει. Και ελπίζω να τα πείτε στους συναδέλφους στο ΕΚΟΦΗΝ αυτό, που δεν κάνανε τίποτα στις προτάσεις τους βρήκαν ένα σύστημα για να ξεφύγουν από τη χρηματοοικονομική εποπτεία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντάνι Κονβέντιτ από τους Πρασίνους. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα πάω προς την ίδια κατεύθυνση που πήγε και ο Γκί Φερχόσταθ. Είναι προφανές. Τέσσερις μέρες παραπέαμε κάναμε, μήνες κάναμε λάθη και οδηγηθήκαμε στην κερδοσκοπία. Τουλάχιστον οι υπεύθυνοι από το Συμβούλιο ας το πούνε. Ας πούνε ότι σφάλαμε. Εμείς, δικό μας το λάθος. Η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαρκοζή, δεν ξέρω εγώ πώς τους λένε και δεν ξέρω τι κάνουν κατά τα άλλα στη ζωή τους. Όλοι το διαβάσανε στις εφημερίδες ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει αμέσως. Δεύτερο. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση Παπανδρέου, αυτό είναι κάτι το αδύνατο σχεδόν. Ζητάω λοιπόν από το ΕΚΟΦΗΝ, από τους ε, ηγέτες κατών και κυβερνήσεων να σκεφτούν ότι αυτοί στις χώρες τους είναι αδύνατο να κάνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Για να μεταρρυθμίσει τι ε, συντάξει η Γαλλία πόσα χρόνια χρειάζεται, η Γερμανία. Και τώρα ζητάμε από τον Παπαδρέο σε τρει μήνες να τα αλλάξει όλα. Μα τρελαθήκατε. Και απόδειξη, να τι έγινε στην Ελλάδα δεν δίνουμε στην Ελλάδα και στον κύριο Παπανδρέου το χρόνο για να μπορέσει να πετύχει συνένεση στην Ελλάδα, για να πετύχει συνένεση εκεί. Δεν υπάρχει ε, συμφωνία. Ο καθένας θέλει το δικό του στην Ελλάδα. Είναι κρίμα. Η συλλογική ευθύνη μετά από δεκάδες χρόνια διαφθοράς ε, ή άλλο πολιτικό στην Ελλάδα δεν μπορεί, δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η συνοχή από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δεν γίνεται με διατάγματα. Και στην Ισπανία θα δείτε αν έχετε το ίδιο πρόβλημα τι θα γίνει. Ή στην Πορτογαλία, αν προκύψουν τέτοια προβλήματα, τι θα γίνει στην Πορτογαλία. Κύριε Μπαρόσο, κάτι ξέρετε. Έχασε με αυτόν τον τρόπο τι εκλογέ. Όχι, α, δεν έχασε ποτέ εκλογέ ο κύριο Μπαρόσο. Καλά. Τι εννοώ. Εννοώ ότι εμεί πρέπει να έχουμε το αίσθημα τη ευθύνη υψηλά. Δεν μπορούμε να ζητάμε τα αδύνατα. Πριν από λίγο καιρό ακούγαμε I want to make money on the back of the Greece. Αυτά ακούμε. Βέβαια, όταν 1,5 με 3% εμείς δανειζόμαστε και δίνουμε με 3,5 5 ε, ή 6% τα δανείζουμε στην Ελλάδα, ε, προφανώς και κερδίζουμε εις βάρος της Ελλάδας, στην πλάτη της. Η Ελλάδα, συγγνώμη, η Ευρώπη μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και είπε ο κύριος Φερχόφσταθ, μίλησε για ένα Ευρωπαϊκό Νομισμό Ταμείο, για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για Ευρωπαϊκό Δανεισμό να αλλάξουμε τις συνθήκες. Ε, ναι, συνάδελφοι, εδώ, μέσα σε αυτό το χώρο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλία για να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Μην περιμένουμε το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να αποφασίσει το Συμβούλιο. Εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία. Μια κοινή πρωτοβουλία εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αλλάξουμε τις συνθήκε ώστε επιτέλους να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει την κερδοσκοπία. Μπορούμε να το κάνουμε. Yes, we can. Ας το κάνουμε. Και τώρα, κάτι άλλο. Για τόσα γίνονται στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βάλει τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης μέσα για να μετρήσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Και ζητάω από το Συμβούλιο να πει στο Διεθνές Μεσονατικό Ταμείο να βάλει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να δει τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί πρόκειται για ανθρώπου. γιατί πρόκειται για προβλήματα απασχόληση. Είναι μισθωτή εκεί. Και δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά τα οποία πρέπει να υπαγορεύουν το τι θα γίνει, αλλά και το διεθνέ Γραφείο Εργασίας ή η Γενική Διεύθυνση απασχόληση. Θα πρέπει μαζί να φροντίσουν να διορθώσουν την τρέλα που έχει πιάσει για την διευθέτηση των δημοσιονομικών. Και κάτι τελευταίο υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουμε τον ελληνικό προπολογισμό. Απλά να αναλάβουμε πρωτοβουλία ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αφοπλισμό στην περιοχή. Δηλαδή, μια πολιτική πρωτοβουλία Ελλάδα, Τουρκία, αφοπλισμός. Δηλαδή, μια πολιτική πρωτοβουλία ώστε τα ελληνικά, τα τουρκικά στρατεύματα, διορθώνω μιλητής, να αποσυρθούν από την Κύπρο να έχουμε αφοπλισμό. Μα είναι υποκριτικό τους τελευταίους μήνες η Γαλλία πούλησε έξι φρεγάτες στην Ελλάδα για 2,5 δις, ελικόπτερα για πάνω από 300 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ναι, η κατασκοπία μου βέβαια δεν μου επιτρέπει να πω ακριβώς τι εξοπλισμό αγόρασε η Ελλάδα. Έπειτα η Γερμανία υποβρύχια, έξι υποβρύχια θα πουλήσει το αποφάσισε πριν από λίγους μήνες στην Ελλάδα. 6 δισεκατομμύρια. Μα είναι υποκριτικό. Τους δίνουμε χρήματα για να αγοράζουν όπλα από εμά. Ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει έκθεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για όλες τις πωλήσει όπλων από την Ευρώπη στην Ελλάδα και την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον υπάρχει διαφάνεια. Να ξέρουμε. Αν θέλαμε να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα ας επιτρέψουμε στην Ελλάδα να χαίρει της ακεραιότητες της εδαφικής της ακεραιότητας Είναι τρελό αυτό που γίνεται με τα στρατεύματα. Με 11 εκατομμύρια κατοίκους έχει 100.000 στρατό. Ας είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν είναι δυνατόν. Και αντί να τα βάζουμε με τους μισθούς κάποιου που βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα. Ας είμαστε λίγο δίκαιοι. Ευχαριστώ από την ομάδα των ε, ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Ντέρκ Γιάνγκ Έπινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Εγώ είμαι αντιπαναστάτης γεννημένο και δεν θα εκφραστώ με τόσο πάθο όσο ο κύριος Μπέντιτ. Και τώρα κατάλαβα το 68 γιατί ήταν τέτοιο ήρωας. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι και τον έβλεπα στην τηλεόραση. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη. Ε, ε, ε, ρωτάνε οι συνταξιούχοι, οι αποταμιευτές, πού πάνε τα λεφτά τους. Γιατί είναι θεμητό αυτό να το ρωτάνε. 110 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Μιλήσατε για 35 δισεκατομμύρια, μετά 60, μετά 110 κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Τεράστιο πακέτο. Και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της. Στα 53 βγαίνουν στη σύνταξη. Και ποιος δεν θα το ζήλαβε αυτό. Και βέβαια τώρα έχουμε απεργίες, εξεγέρσεις, επεισόδια. Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι δικό μας πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Αθήνα, κύριε Κονμπέντιτ, αφορά τους ε, Ολλανδούς, τους Φλαμανδούς, τους Γερμανούς, τους πάντες. Και παραμένει ο κίνδυνος μετάδοσης. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να του είχαμε βγάλει από την Ευρωζώνη του Έλληνε όταν διαπιστώθηκαν αυτέ οι ατασταλίε και τα προβλήματα. Του αφήσαμε και θα πρέπει να δούμε το ε, σύμφωνο σταθερότητας και τους κανόνες. Ποια είναι η σταθερότητα, πού είναι η οικονομική ανάπτυξη. Ε, ισχυρή εποπτεία, το ξέρω. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο θαραλέα. Μεγαλύτερη εποπτεία στην εφαρμογή των κανόνων. Δεν συνέβησαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Κατά την άποψή μου όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία εξόδου από την Ευρωζώνη για μια χώρα που δεν αντέχει να είναι πλέον στο ευρώ. Τι να κάνουμε. Δεν λέω να τους βγάλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη. Και θα πρέπει να υπάρχει αυτό το θάρρος. Να κάνει ειδικό του νόμισμα ξανά το κράτος, να κάνει και υποτίμηση και να μπορεί να αρθοποδεί ξανά. Να παραμένει με τη Λισαβόνα ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της Ευρωζώνης. Μα τώρα μιλάμε για πιο στενή ένωση. Ever Closer Union. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Ισχύουν τώρα. Με, έχουμε και ε, χαμηλή ανάπτυξη και ασταθές ευρώ. Και πού είναι αυτή η θεωρία. Έχουμε καταστήσει ο ε, τους φορολογούμενους της χώρας μας και ο κόσμος ανησυχεί. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς ε, το λόγο έχει ο Πρόεδρος Μπίσκι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και βέβαια η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια. Αλλά η λεγόμενη δράση διάσωσης έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γαλλία, Γερμανία, μεγάλες δυνάμεις πήραν την απόφαση για το πακέτο βοήθειας και ε, μεγάλες καθυστερήσεις που κοστίζουν ακριβά. Οι χρηματαγορές εδώ και χρόνια έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους, απορριθμίζονται συνεχώς και τώρα όλοι εκπλησόμαστε ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Και ποιο θα πληρώσει την ύφη? Οι εργαζόμενοι, οι άνδρες και οι γυναίκες, ο Κοσμάκης, όχι οι τράπεζες, δεν θέτουμε ενώπιον των ευθυνών τους και πάλι οι φορολογούμενοι θα την πληρώσουν. Και θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, το κεφάλι τους, ε, για να τους καρατομήσουν. Και πάλι περικοπές μισών, με επιταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και δημιουργείται και η εντύπωση, η εικόνα ότι είναι δημοκρατική διαδικασία. Στο Μεξικό με την πετρελογική κοιλίδα εφαρμόζεται, απαιτείται η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Όποιος ψάχνει λεφτά ή όποιος ψάχνει χρυσό θα πρέπει να ξέρει ότι θα υφίσταται και τις ζημίες. Οι τράπεζες, τουλάχιστον στη Γερμανία προς το παρόν, δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν ούτε καν τα χρέη που ανέλαβαν να καλύψουν. Και χαροπά κερδοσκοπούσαν εις βάρος του ευρώ. Και, και το δέχομαι και συνεχίζουν να το κάνουν. Παρόλο που εδώ και καιρό ζητούμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Προτάσεις. Τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν. Απαγόρευση εμπορίου των παραγόγων και των χρεογράφων. Ε, φόρος, τέλος στις συναλλαγές φορολόγηση των πόνους. Τέλος, ε, ε, διανόμου να επιβάλλεται στις συναλλαγές. Όλα αυτά υπάρχουν ως προτάσεις. Βεβαίως θα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει τα δικά της καθήκοντα. Όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει και η Ελλάδα να φορολογεί τον πλούτο, να καταπολεμά τη διαφθορά και να μειώνει τις εξοπλιστικές της δαπάνες πολύ επιστικά τα όσα είπε προηγουμένως ο Κον Μπέντιτ και δεν χρειάζεται να σας αναφέρω άλλα στοιχεία. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Μπορώ να καταλαβαίνω τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους στην Αθήνα και διαμαρτύρεται. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η βία. Και συμφωνώ κι εγώ και προσθέτω τη φωνή μου και στα συλληπιτήρια των ε, οικογενειών των θυμάτων γιατί η βία έχει το αντίθετο αποτέλεσμα ε, από εκείνο που θέλουν οι άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά και ειλικρινά. Παρακαλώ, όχι βία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εξ ονόματος της ε, Ομάδας Ελευθερίας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαλαβράκος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, προσπαθούμε να εξορίσουμε τους αριθμούς και είναι γνωστό ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί δυστυχούν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και τους αριθμούς να ισορροπήσουμε και την ευτυχία των ανθρώπων να δώσουμε και να διατηρήσουμε. Αποτέλεσμα αυτής της ανορθόδοξης συμπεριφοράς ήταν ότι σήμερα στην Ελλάδα θρυνούμε τρία θέματα το θάνατο τριών εργαζομένων από την επιθετική διαμαρτυρία άλλων εργαζομένων σε όλη την ευρώπη σήμερα η οικονομική κρίση που μας ήρθε από την άλλη πλευρά του ατλαντικού και τίνει να γίνει χειρότερη σε μας ε, έχει τίνει να απαξιώσει την πολιτική ζωή και τους πολιτικούς. Στην Ελλάδα υπάρχει στα λαϊκά στρώματα μια πάρα πολύ κακή διάθεση απέναντι των πολιτικών. Έχουμε 300 στην Ελληνική Βουλή. Ακούω στον παλμό της ελληνικής κοινωνίας δεν δηλαδή είναι να κρεμάσουμε τους 300. Είναι επικίνδυνα πράγματα. Διαβάζω τα ίδια πράγματα και την ίδια απαξίωση της πολιτικής η οποία έχει έρθει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όλοι το ξέρουμε και όλοι επίσης ξέρουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη δημοκρατία. Με τα δεδομένα και με τις σκέψεις αυτές, διότι δεν μπορώ, δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ περισσότερο, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι οι ηγέτες μεθαύριο θα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα και στην κατεύθυνση μιας μονιμότερης λύσης και για περισσότερα κράτη. Η Ελλάδα είναι το ένα. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν και άλλα κράτη και μέλη της Ευρωζώνης και μη μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα που θα έρθουν εντονότερα τους προσεχούς μήνες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας διάκοψα γιατί είστε Έλληνας και ήταν πολύ σημαντικά τα λόγια σας για όλους μας. Και τώρα ο κύριος Μπάρι Μάτλενερ από τους μη εγγεγραμμένους. 1,5 λεπτό. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το Φερχόφστατ και το Σούλτς που δεν είναι εδώ, αλλά παρεμβρίσκεται η ομάδα του, σοσιαλιστές. Γιατί είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα. Τώρα δείχνουν υποτίθεται αλληλεγγύη. Χρειάζεται αλληλεγγύη, αλλά θυμηθείτε ότι η Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι καθαρός αποδέκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα ερχόμαστε τόσα χρόνια μετά να διεργνύουμε τα, τα ημάτια μας. Πού ήταν η κριτική στο παρελθόν. Και τώρα, ορίστε, ε, ε, είμαστε πρωτετελεσμένων γεγονότων. Ακούσουμε και στην Ισπανία. Δύο, ε, εκατομμύρια λάθρομετανάστευση νομιμοποίησε τα τελευταία 15 χρόνια και τα βρίσκατε όλα αυτά θαυμάσια και τώρα έχουν 20% ενεργεία. Και μετά η Πορτογαλία. Εκεί κυβερνάνε οι σοσιαλιστέ που τους υποστηρίζετε τόσα χρόνια με ευρωπαϊκά χρήματα. Και κάναμε τώρα αυτή την τρύπα στο νερό και τώρα θα πληρώσουμε εμείς την ύφη και οι πολίτες μας. Κανονικά έσχο, έπρεπε να ντρέπεστε. Τώρα λέτε θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Δεν αντέχουν την Ευρωζώνη να ξαναφέρουν τη δραχμή. Και αν συμβεί το ίδιο στην Ισπανία, να φέρουν και την πεσέτα ξανά και το εσκούδο γιατί αυτή η Ευρώπη είναι στρεβλή Ευρώπη και οι Βορειοευρωπαίοι αρνούνται να πληρώσουν τα δικά σας λάθη και τις ε, σοσιαλιστικές ε, επιπόλαιες κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες. Ε, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, γεμάτο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, καθαροί αποδέκτες των χρημάτων, ε, οργιάζει η λαθρομετανάστευση και εσείς με σταυρωμένα τα χέρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Για διαδικαστικό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο, αλλά επειδή αναγνωρίσατε τον κύριο Σαλαβράκο και ω Έλληνα παρόντα, θέλω να αναφερθώ σε ένα πράγμα το οποίο είπε. Ανέφερε ότι τρει άνθρωποι σήμερα σκοτώθηκαν στην Αθήνα, τρει εργαζόμενοι, από τρει άλλου εργαζόμενου. Αυτό είναι απολύτω λάθο. Σκοτώθηκαν από δολοφόνου, από εγκληματίε. Οι εργαζόμενοι στην Αθήνα σήμερα είχαν μια ειρηνική, ειρηνική μεγάλη πορεία δεν σκότωσαν κανέναν και καταδικάστηκαν αυτοί οι εγκληματίες από τον πρωθυπουργό τον γιώργο παπανδρέου και από όλα τα πολιτικά κόμματα στη βουλή πριν από λίγη ώρα. είναι πολύ μεγάλο λάθος και επικίνδυνο να υπάρχει σύγχυση μεταξύ ειρηνικών διαδηλώσεων και εγκληματικών πράξεων όπως αυτές που συνέβηκαν στην αθήνα καταδικάζονται από όλους και δεν εκφράζουν ούτε τον ελληνικό εργαζόμενο ούτε την πεποίθηση όλων ότι ενωμένοι πατριωτικά θα βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κρίση. ευχαριστώ. E, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρινίδη, που μας δώσατε τις επεξηγήσεις αυτές. Δεν θέλω να μπούμε σε συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά θέλω να επαναλάβω ότι όλοι οι ευρωβουλευτές εκφράζουμε και εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπής δίχω άλλως Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας. Ξέρουμε ότι την ευθύνη την έχουν και οι δύο πλευρές. Εγώ έχω περάσει και εγώ προσωπικά από τέτοιες καταστάσεις. Ήμουν ενεργό μέλος συνδικάτου και Πρωθυπουργό κατά το παρελθόν και έτσι μπορώ να καταλάβω την κατάσταση στην Ελλάδα. Εννοείται ότι σκεφτόμαστε πολύ τις οικογένειες των θυμάτων. Χρέος μας είναι να μην τους ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Τώρα το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο κύριος Λόπες Γαρίγα, εκ